Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Άρχεται η συνεδρίαση. Ε, το πρώτο θέμα είναι η έκθεση του κύριου Βενσάν Πεγιό με θέμα την Ένωση για τη Μεσόγειο. Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής για τέσσερα λεπτά, παρακαλώ. Mm. Euh, euh, Καταρχάς ευχαριστώ θερμά όλους του συναδέλφους που συμμετέχουν στην εργασία αυτή που είναι πραγματικά συλλογική. Έχουμε 28 συμβιβασμούς και που μάλιστα δεν ε, αποδυνάμωσαν καθόλου την έκθεση αλλά την εμπλούτησαν. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά την Μαριέτα Γιαννάκου από το ΕΛΚ, τον Ιβο Βάγκελ για τους φιλελεύθερους, την Ελένη Φλότρα και τον εισηγητή της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου κυρία Αντεσαρνές και της βιομηχανικής την κυρία Σαβέλα. Για μας το σημαντικότερο είναι να καταλάβουν όλοι ότι εδώ υπάρχει ένα στρατηγικό συμφέρον της Ευρώπης δηλαδή δεν χρειάζεται απλώς να φανεί ότι ο Νότος μας χρειάζεται, αλλά ότι και εμείς χρειαζόμαστε τον Νότο, ιδίως σε τέτοιες στιγμές κρίσεων. Και αν θέλουμε μακροπρόθεσμα να έχουμε κάποια όραμα, κάποια βιώσιμη ανάπτυξη σε έναν κόσμο πολυπολικό, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε και τον Νότο μας. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να δεσμευτεί να κάνει την Ένωση για τη Μεσόγειο έναν χώρο ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας για 800 εκατομμύρια ανθρώπους ε, και να το καταστήσει αυτό προτεραιότητα. Η κοινή αυτή θέληση μας επέτρεψε να ενώσουμε τις προσπάθειές μας αντιμετωπίζοντας οικονομικά, δημογραφικά, γεωπολιτικά προβλήματα που πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία οι δύο όχθες της Μεσογείου. Είναι για μας θέμα και πολιτιστικό και πολιτισμικό. Το Κοινοβούλιο γνώριζε πόσο δύσκολη θα ήταν η εφαρμογή των σχεδίων αυτών για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Δεν αποφύγαμε τις διαμάχες, ούτε θελήσαμε να τις κρύψουμε, που υπάρχουν μεταξύ των χωρών του Νότου, αλλά θελήσαμε να δείξουμε ότι το όραμα της Ένωσης και τα συγκεκριμένα της προγράμματα, η ισότητα βορρά και νότου στην εκπροσώπηση και η δυνατότητα κοινών συναντριάσεων μεταξύ ας πούμε Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι η σωστή μέθοδος για να μπορέσει και η Ένωση να συμβάλλει στην επίλυση τέτοιων διαμαχών. Εξάλλου η Ένωση για τη Μεσόγειο δεν θέλησε να λύσει ταυτόχρονα όλα τα προβλήματα και να θίξει όλους τους στόχους ταυτόχρονα, αλλά να μιλήσει με συγκεκριμένη γλώσσα. Θα ήθελα λοιπόν η δεύτερη διάσκεψη της Βαρκελόνης του 7 Ιουνίου να δείξουμε εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ότι χρειάζεται μεγαλύτερη δέσμευση ώστε να πετύχει η διάσκεψη αυτή. Και μιλήσαμε για τους δρόμους που μας ανοίγονται. Δηλαδή πρέπει πρώτον να βγουν από τη μέση διάφοροι φραγμοί μεταξύ των οποίων τα δημοσιονομικά. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να υπάρξει μια χρηματική δέσμευση της Ένωσης αντίστοιχη με το μέγεθος των προβλημάτων και στις δημοσιονομικές προοπτικές 14 με 20 η δέσμευση της Ένωσης να αυξηθεί πολύ για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που υπάρχουν. Χρειαζόμαστε βελτίωση του οικονομικού και νομοθετικού περιβάλλοντος ώστε η περιφερειακή διάσταση να ληφθεί πλήρως υπόψη και πέρα από αυτά να δημιουργηθούν και νέες πολιτικές συνθήκες και γι' αυτό επιμείναμε τόσο πολύ στη, στα πολιτιστικά, στα ανθρώπινα δικαιώματα και Καταλήγω εδώ κύριε Πρόεδρε δηλώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει όραμα μακροπρόθεσμο και να αναλάβει τις ευθύνες της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πεγιόν. Και τώρα έχει το λόγο ο Επίτροπος κύριε Φίλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε, ε, κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ιδιαίτερη χαρά ε, σήμερα για μένα ευκαιρία που έχω να μιλώ ενώπιό σας για την Ένωση για τη Μεσόγειο και την έκθεση του αξιότιμου βουλευτού κυρίου Βενσάν Πέγιο. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη η έκθεση αυτή του Κοινοβουλίου γιατί αναφέρεται ακριβώς στις προκλήσεις κλειδιά ε, που θα αντιμετωπίσει τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ένωση για τη Μεσόγειο. Ε, θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ απολύτως ε, κύριε εισηγητά, τα είπατε στην εισαγωγή σας. Τώρα έχει τεθεί πλέον σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ενισχυμένη θεσμική ταυτότητα και μπορεί καλύτερα να ε, δράση και για τον υπόλοιπο κόσμο με εξωστρέφεια πλέον. Οι ε, κυβερνήσεις ε, της Ένωσης για τη Μεσόγειο επίσης έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες. Η πολιτική γειτονία επίσης αλλάζει τα δεδομένα. Από το 2004 έχουν αρχίσει πολιτικές επαφές και η συνεργασία έχει ενταθεί. Έχει διπλασιαστεί το εμπόριο σχεδόν ε, με την απελευθέρωση και ε, τη σύγκληση των οικονομιών και η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση διαδραματίζει πολύ σημαντικό οικονομικό ρόλο. Η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αλλά και ως πηγή διμερούς συνεργασίας δημερού συνεργασία ορισμένων κρατών μελών της Ένωσης με ε, χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη ολοκλήρωση, ευρωμεσογειακή ολοκλήρωση για να μπορέσουμε να ε, οδηγηθούμε στην απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη, στι επενδύσει, και αυτό να είναι προ όφελο όλων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών τη Μεσογείου. Έτσι ε, θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με ε, κοινέ αξίες. Έχουμε ε, συμφωνίες ε, με τις χώρες αυτές που έχουν πάρα πολύ νέο πληθυσμό. Ε, Ένωση για τη Μεσόγειο ε, ξεκίνησε στο Παρίσι το 2008 και αυτό έδωσε ε, μια νέα όθηση στην ευρωμεσογειακή συνεργασία. Για κοινή ευθύνη, για κοινή προσπάθεια, με ένα σύστημα ε, συμπροεδρίας που εστιάζεται σε συγκεκριμένα προγράμματα και μια τεχνική γραμματεία για να προωθήσει την περιφερειακή ολοκλήρωση. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η εφαρμογή επιβραδύθηκε από την αύξηση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ο πρόοδος έχει επιτευχθεί ε, με την ε, συζητήσει της Παλαιστινιακή Αρχής με την Ισραηλινή κυβέρνηση μπορούμε να πούμε ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι μπορεί ε, τελικά να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη συνεργασία στην περιοχή. Είναι τεράστιες οι παγκόσμιες προκλήσεις, ε, όπως ε, η ε, διεθνής οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή ασφάλεια. Η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει ακριβώς να αντιμετωπίσει και την πολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Να αρχίσει η λειτουργία της γραμματείας και να καταγραφεί η πρόοδος που έχει γίνει από τον Ιούλιο του 2008 μέχρι σήμερα. Είναι ευκαιρία λοιπόν συλλογικά να διατρανώσουμε και πάλι την προσήλωσή μας και την πολιτική μας βούληση για να δημιουργήσουμε ένα χώρο ασφάλειας, ε, ειρήνης και συνεργασίας στη Μεσόγειο και για να γίνει αυτό θα πρέπει ε, οι εταίροι ακριβώς να ασχοληθούν και να διαφερθούν με την οικονομική ανάπτυξη επιτόπου, δηλαδή έργα, ε, ε, θέσεις απασχόλησης και οικονομική μεγέθηση. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή η Μεσόγειος και η νέα γενιά ζητάει καλύτερες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Ζητούν περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη δημοκρατική εκπροσώπηση. Ε, ε, για ε, μεγαλύτερη και καλύτερη μόρφωση, δυνατότητα μετακίνησης, ταξίδια να κάνουν, γνωρίζουν τον κόσμο και θα πρέπει να υποφελούνται από την κοινή μας δράση. Εάν έχουμε συγκεκριμένα έργα, πρόσβαση σε ενέργεια, σε νερό, σε τροφή, πολιτική προστασία, αυτό είναι ακριβώς προς όφελος των λαών των χωρών αυτών. Η Ένωση της Μεσογείου έχει ε, ως σκοπό να βοηθήσει ε, τον κόσμο, επιχειρηματίες, ΜΚΟ, πανεπιστήμια και κυρίως νέους ανθρώπους που είναι ε, στην πρωτοπορία της συνεργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και μέσα από την πλήρη συμμετοχή και των εκλεγμένων εκπροσώπων των λαών. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι βαθύτερα πεπισμένη ότι χρειάζεται μια ισχυρή και παλόμενη κοινοβουλευτική διάσταση για να βοηθήσει. Εξού και η ε, Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση θα πρέπει να ενισχυθεί, να εδρεωθεί ε, και να συνεργαστεί με άλλα θεσμικά όργανα και σώματα τη συνεργασίας. Εμείς θέλουμε να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μεσόγειο συγγνώμη, και θα κρυθεί από τα πραγμένα και από τα αποτελέσματα για την περιφέρεια. Ε, ε λεωφόροι, διασυνδέσεις ε, στην ενέργεια, λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη ε, το ηλιακό επίσης πρόγραμμα ε, για τη Μεσόγειο είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για ε, επενδύσεις, θέσει απασχόλησης και ενισχυμένη συνεργασία. Εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό αυτό, χρειαζόμαστε και τον ιδιωτικό τομέα και σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα χέρι με χέρι. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένας καταλήτης και ο καταλήτης αυτό είναι η γραμματεία για την Ένωση της Μεσογείου μετά από πολλούς μήνες ε, σκληρής δουλειάς επιτέλους καταφέραμε να εγκρίνουμε ε, το καθεστώς της γραμματείας, να ορίσουμε γενικό γραμματέα και να εγκρίνουμε προσωρινό λειτουργικό προϋπολογισμό. Στην καρδιά των σχέσεών μας με τους εταίρους μας στη Μεσόγειο είναι η επιθυμία μας να προωθήσουμε την ασφάλεια, την ε, ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Αλλά επίσης είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι συμμετέχουμε σε ένα σχέδιο ακόμα πιο φιλόδοξο. Να είναι περιοχή ειρηνική και να έχουμε κοινέ αξίες και αρχές. Είμαι βέβαιος ότι από κοινού και με τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτύχουμε και με τη μεγάλη συνεργασία της Ευρωμεσογειακής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. You, Commissioner. Now our next Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Ντεσάρνες. Mm. Βεβαίω, ε, η διαδικασία τη Βαρκελόνη είναι αβέβαιη και σίγουρα ε, καθυστερεί λόγω της, ε, σύγκρουση ε, της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινή, αλλά και σίγουρα βοηθάει στο να βελτιωθεί ο διάλογο ανάμεσα στι δύο όχθε τη Μεσογείου. Χρειάζονται οικονομικέ και οι πολιτιστικές συναλλαγές. Χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για το μέλλον που θα κινητοποιεί την ενέργεια όλων των κρατών. Μέσα σε αυτό το πνεύμα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε τι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και η Κομισιόν ε, θα πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να ενισχύσει το ρόλο της ως επενδυτή ε, Επίση, να ενισχύσει τη διαδικασία τη ε, απελευθέρωση όταν γίνονται οι συμφωνίε νέα γενναία. Τέλο, η συμφωνία του Αγαδίρ θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη ανταλλαγή, προώθηση μάλλον των συναλλαγών νότου-νότου. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί επίση η διατροφική ασφάλεια και όλοι το γνωρίζουμε πω το θέμα τη ενέργεια είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν θα πρέπει να γίνουν ενέργειε προ το συμφέρον αυτών των χωρών ώστε να συμβάλλουμε στις δικαι... στην κάλυψη των δικών του αναγκών παρά τι δυσκολίε και επειδή ακριβώ υπάρχουν αυτέ τι δυσκολίε. Έχω 1,5 λεπτό, υπάρχει λάθο εκεί στον πίνακα. Λοιπόν, και παρά τις δυσκολίες και μάλλον λόγω των δυσκολιών θα πρέπει να ε, δοθεί νέα όθηση στις... Ναι, με ευρωμεσογειακή ε, ε, συνέλευση. Ευχαριστώ, κυρία Τζαβέλα. Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεσή μας για την ευρωμεσογειακή αγορά βεβαιωθήκαμε ότι εισηγούμαστε την διατήρηση και ανάπτυξη των βασικών υποδομών που συνθέτουν μια οικονομία ενιαία και συνεκτική και είναι ενδιαφέρον ότι τώρα με την οικονομική κρίση η συγκυρία επιδεικνύει πολύ ε, εμφανώς ότι υπάρχει μια συνοχή και κοινά χαρακτηριστικά στο νότο. αυτό ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας για κάποιες μελλοντικές εξελίξεις. ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έκθεσή μου στο lng το οποίο πολύ βραχυπρόθεσμα μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο οικονομική δύναμη για την οικονομία της ευρωμεσογειακής αγοράς όχι μόνο για προμήθεια αλλά και για πώληση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μια άλλη ε, πηγή ε, οικονομίας για την ευρωμεσόγειο οι οποίες όμως είναι πιο βραχυπρόθεσμες. μια ε, παρατήρηση η στρατηγική και η πολιτική της Ένωσης όσον αφορά ε, την ε, ενέργεια για τη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη. Έχουμε, κύριε Επίτροπε, μεγάλη αδυναμία mm-hmm. στην πολιτική και στρατηγική για την mm-hmm. ενέργεια mm-hmm. στο νότο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ακολουθούν οι πολιτικές ομάδες εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η κυρία Γιαννάκου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Βενσάν Πεγιόν καθώς και τις εισηγήτριες από τις άλλες επιτροπές, την κυρία Ντεσαρνές και την κυρία Τζαβέλα για την εισήγησή τους. Η έκθεση για την Ένωση για τη Μεσόγειο είναι σημαντική γιατί επικεντρώνεται σε άμεσους και μετρήσιμους στόχους. Τα αποτελέσματά τους μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένα αφού το Κοινοβούλιο ζητά μέσω της έκθεσης ε, να δοθεί συγκεκριμένος προϋπολογισμός μέσω των δημοσιονομικών προοπτικών να βοηθηθεί η γραμματεία της ένωσης η οποία βρίσκεται στη Βαρκελόνη και βεβαίως οι διάφορες συγκρούσεις που υπάρχουν να μην μπορούν να επηρεάσουν τον καθαυτό στόχο της ένωσης που είναι η ανάπτυξη η προσπάθεια για τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα πολιτιστικές ανταλλαγές τα ζητήματα της ενέργειας και ό,τι μπορεί να συνδέσει στη λεκάνη της μεσογείου τους λαούς οι οποίοι είναι εκεί. Βέβαια σήμερα εδώ κύριε Πρόεδρε λείπει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο και η Ισπανική Προεδρία η οποία υποθέτω ότι έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μεσογειακή Ένωση και πρέπει να σημειώσω ότι αυτό με εκπλήσει γιατί το Συμβούλιο θα έπρεπε να ακούσει όσα είπε ο εισηγητής και οι συνεισηγήτριες αλλά και όσα τονίζονται εδώ ότι δηλαδή είναι μια προσπάθεια είναι μια υπέρβαση των συγκεκριμένων δυσκολιών βάσει των οποίων τα προγράμματα δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν όπως πρέπει. η, διαμάχη μεταξύ παλαιστινίων και ισραηλινών βεβαίως δεν λύεται μέσω της ένωσης για τη μεσόγειο αλλά οπωσδήποτε η ύπαρξη αξιωματούχων στη γραμματεία δίνει μια ελπίδα ότι δεν θα υπάρχει η πίεση των συγκρούσεων στην προσπάθειά μας ε, να προχωρήσει η ένωση για τη μεσόγειο με τα κριτήρια που ελέγχθησαν προηγουμένως. κύριε πρόεδρε έχει ιδιαίτερη σημασία για την ένωση επίσης να δώσει ένα μήνυμα για τη δημοκρατική εξέλιξη την ισότητα ανδρών και γυναικών και την προσπάθεια για κοινωνία πολιτών και στις χώρες της βορείου αφρικής. σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ο κύριος ε, Ομπιόλ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από την έκθεση αυτή και συγχαίρω επ' ευκαιρία το Βενσάν σάμπεγιον τον εισηγητή μας, είναι ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πολύ ακριβής η έκθεση. Μακάρι η ακρίβεια αυτή της εκθέσεως να ε, επεκτηνόταν και στην πραγματικότητα. Ε, για την οποία αναφέρεται, στην οποία αναφέρεται ε, στην Ένωση για τη Μεσόγειο, γιατί το ελάχιστο που μπορεί κανείς να πει είναι ότι στην Ένωση για τη Μεσόγειο επικρατούν πολύ μεγάλες ασάφειες και θα συνδυάσουν οι ηγέτες, ελπίζουμε τουλάχιστον στις 7 Ιουνίου στη Βαρκελόνη, ε, καλά θα κάνουν να ακολουθήσουν τις συγκεκριμένες και ακριβείς προτεραιότητες που αναφέρει η έκθεση Πεγιό. Πρώτον, για ε, το πολιτικό γίγνεσθε. Η Ένωση για τη Μεσόγειο δεν μπορεί να παραμείνει σε ομοιρία και σε παράλυση από τη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί και να το αγνοήσει αυτό το γεγονός. Θα πρέπει ε, στο μέτρο του δυνατού να φέρει και θετικά στοιχεία για την επίλυση της διένεξης αυτής. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι καλά τα έργα, να γίνονται επαγγελματικά και με ευφυΐα και να τα προωθούμε. Και τρίτον, θα πρέπει να βρούμε τους απαραίτητους πόρους και τους οικονομικούς ε, και επαρκείς όμως. Και τέταρτον, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια καλή σχέση χωρίς εμπόδια ε, και χωρίς ε, προσκόμματα με συνεργασία με τις χώρες της Μεσογείου στις δομές ε, της Ένωσης και τη Μεσόγειο. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά στοιχεία, οι τέσσερις βασικές προκλήσεις και εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε σαφήνεια και δέσμευση. Και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι ένα καλό εργαλείο, είναι ένα καλό φύλλο πορείας για να φτάσουμε στη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ κύριος Βάικελ από τους φιλελευθερού Δύο μισή λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε μαζί του με αποτέλεσμα την έκθεση που έχουμε μπροστά μας. Ελπίζω να αποβεί ενδιαφέρουσα και για άλλους, όχι μόνο για μας, τους συντάκτες. αναφέρεται σε μια περιοχή που υπήρξε δυναμικό κέντρο της πνευματικής και οικονομικής ζωής όλη, καθ' όλη την ανθρώπινη ιστορία. Δυστυχώς όμως σήμερα παραμένει πηγή πολλών προβλημάτων που θα θέλαμε όλα να λυθούν. Η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν προχωράει τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε. Θα θέλαμε να δημιουργηθεί γραμματεία στη Βαρκελόνη και να γίνει πρόοδος για την επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων που έχουν καθοριστεί. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμή πολιτικά θέματα όπως το Παλαιστινιακό και το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Πράγμα που, πράγματα που εμποδίζουν την πρόοδο και χρειάζεται περισσότερη ανοχή, διάλογος και εμπιστοσύνη το ευρωπαϊκό όραμα μπορεί να συμβάλλει θετικά ως προς αυτό και με χαρά διαπιστώνουμε ότι γίνεται αποδεκτό από όλους τους παράγοντες εκεί. Τέλος θα ήθελα να προσθέσω ότι πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τη σημασία των μελλοντικών γενεών να τη στηρίξουμε από την πλευρά της Ένωσης να οργανώσουμε ανταλλαγές φοιτητών, πολιτιστικά βήματα, πράγμα το οποίο να αυξήσει ακριβώς την εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής η κυρία Βεναρά Μπατού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ένωση για τη Μεσόγειο δεν ήταν ποτέ τόσο ζωτική για το μέλλον μας όσο σήμερα. προσπαθήσαμε από κοινού μέσα στην έκθεση αυτή να στηρίξουμε διάφορες ε, περιφέρειες της Μεσογείου μας. Πολύ περισσότερο από μια απλή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών πρόκειται για μια ένωση που βασίζεται σε ένα κοινό πολιτισμό τον οποίο συμμερίζονται άνθρωποι που με κοινέ αξίες. Ήθελα να σας ε, μιλήσω για τη βία την οποία υπόκειται ο Παλαιστινιακός λαός, ε, ο οποίος είναι υπό την Ισραηλινή κατοχή, χωρίς εμείς να αναλαμβάνουμε τις ιστορικές μας ευθύνες σε αυτή τη σύγκρουση. Ε, θα πρέπει να, να αγωνιστούμε για την ειρήνη, να αναγνωρίσουμε το Παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με τις διεθνείς νομοθεσίες επί των οποίων βασίζονται και οι δημοκρατίες μας. Την επόμενη εβδομάδα μια επίσημη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα μεταβεί στη Λωρίδα της Γάζας για να καταλάβει γιατί η βοήθεια που στέλνουν οι Ευρωπαίοι στους Παλαιστινίους με εκατοντάδες δηλαδή εκατομμύρια ευρώ δεν φτάνει μέχρι τα σχολεία και τα νοσοκομεία της Γάζας όπου εγώ μετέβη την περασμένη μήνα. Ε, πραγματικά έχω σοκαριστεί, ανησυχώ. Ε, ε μόλις έμαθα πως ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων χωρίς να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής ούτε τους συμπροέδρους τη αντιπροσωπείας αποφάσισε να μην πάει στη Γάζα με την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου μας μετά από τις υποδείξεις της πρεσβείας του Ισραήλ. Mm. Βοηκοτάροντας την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Γάζα, ο πρόεδρος της Επιτροπής μας απαξι... απαξιώνει ολόκληρη το Κοινοβούλιο μας, το οποίο στην έκθεση Γκόλστοκ υποστήριξε πως ε, και καταδίκασε μάλλον το γεγονός πως ο Παλαιστινιακός λαός στις, στις είναι εγκλωβισμένος από τις ε, Ισραηλινές δυνάμεις. Υπό αυτές τις ε, συνθήκες ε, ζητώ την παρέτηση του κύριου Αλμπερτίνη από την Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων διότι δεν εστάθη στο ύψος των απαιτήσεων του ρόλου του και της, του λειτουργήματός του. Επιπλέον, Θα πρέπει να διενεργηθούν εκλογές ώστε να υποστηριχθούν αυτοί που επέλεξαν την οδό των, ε, της αντί την οδό των όπλων. Ε, η, μεταναστευτική μας πολιτική από την άλλη πλευρά δεν είναι αποδεκτή πλέον. Θα πρέπει να επιτρέψουμε την κινητικότητα των πολιτών του Νότου σε σχέση με τη δική μας ε, κινητικότητα στο Νότο. Ας είμαστε πιστοί στα σχέδιά μας και στις αξίες μας. Τα παιδιά μας θα μας είναι ευγνώμονα και θα πρέπει να, να αναγνωριστεί αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάγερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, η Ένωση για τη Μεσόγειο έχει αντικειμενικά εμπόδια. Αυτό που θα ζητούσα εγώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο μας είναι αποφασιστικότητα, πολύ ε, περισσότερο στένος όταν προσπαθούμε να υπερβούμε τα εμπόδια. Τα πρώτα και πιο σημαντικά, υπόθηκαν και από άλλους βουλευτές, είναι οι διενέξεις. Η διενέξη ε, στην Παλαιστίνη απέναντι σε μια στάση της Ισραηλινής κυβέρνησης που συστηματικά παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις λίγες συμφωνίες που έχει υπογράψει του της Ινδιανάπολης με τις επικισμούς, η Δυτική Σαχάρα που είναι και αυτή η διένεξη και βεβαίως και η στρατιωτική κατοχή της Βορείας Κύπρου. Είναι αντικειμενικά εμπόδια αυτά και κανένα όργανο, κανένα θεσμικό όργανο που θέλει να έχει ε, ε, αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει μέχρι να λυθούν αυτές οι διενέξεις. Είναι υπαρκτά εμπόδια. Εμείς από την ομάδα μου ζητούμε μεγαλύτερη δέσμευση, περισσότερη ενέργεια απέναντι σε όλους αυτούς τους φορείς που παραβιάζουν ε, το διεθνές δίκαιο και αυτοί είναι υπεύθυνοι. Ε, επίσης όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις διάφορες ασυμμετρίες που επικρατούν στη Μεσόγειο παντού και κοινωνικές και οικονομικές. Οποιαδήποτε φόρμουλα προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την ασυμμετρία δεν θα πρέπει να επιζητά μόνο το κέρδο και συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Δεν είναι σωστή η κατεύθυνση αυτή. Η σωστή κατεύθυνση είναι να λάβουμε υπόψη μα τι ασυμμετρίε και να προσπαθήσουμε να ε, βρούμε εκείνε τι εμπορικέ συμφωνίε που βασίζονται στη συμπροματικότητα και στην αλληλεγγύη. Διότι πολλέ χώρε από την όχθη της Μεσογείου, αυτή την νότια, ε, είναι σε πλήρη ένδια και σε πλήρη περιθωριοποίηση. Αλλά επιμένω, το βασικό θα ήταν από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση στι διενέξει αυτέ που ε, έχουν εδρεωθεί και διονύζονται, που είναι η Δυτική Σαχάρα και η Παλαιστίνη, να λυθούν. Και στη Δυτική Σαχάρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει απολύτω τίποτα. Όχι μόνο δεν κάνει τίποτα, αλλά ε, αναβαθμίζει και το καθεστώ που έχει το Μαρόκο. Και θέλω να βάλει και το Ισραήλ σε αυτό το καθεστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάγερ. Και τώρα ο κύριος παρακαλώ από την ομάδα του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, οφείλω να συγχαρώ το συντάκτη της έκθεσης των κύριο Πεϊών για την, αξιολόγηση, για την αξιόλογη έκθεση που μας παρουσίασε. Είναι γνωστό ότι η λεκάνη της Μεσογείου είναι ένα σημείο συνάντησης πολλών πολιτισμών αλλά είναι συνάμα μια περιοχή νευραλικής σημασίας και ένα καζάνι που βράζει και μάλιστα βράζει εδώ και πολλά χρόνια. Η κλιματική αλλαγή, η η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση η μετανάστευση και η ρήπαση, η υπεραλίευση η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος είναι κάποια από τα προβλήματα που ταλανίζουν τους ευρωπαίους και μη κατοίκους της μεσογειακής λεκάνης. ιδιαίτερα πρέπει να δοθεί σημασία στο θέμα της λαθρομετανάστευσης στον αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων ε, των χωρών της λεκάνης της μεσογείου ιδιαίτερα της ελλάδας και της ιταλίας που αποτελούν θύρες εισόδου λαθρομεταναστών στην ευρωπαϊκή ένωση. μια καθημερινή μάχη δίδεται στα σύνορα των χωρών αυτών. έμφαση επίσης πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μάλιστα στην αξιοποίηση του μεσογειακού προγράμματος ηλιακής ενέργειας για την οικονομική mm. ανάπτυξη των νοτίων χωρών της μεσογείου. ευχαριστώ πάρα πολύ. Mr. Ο κύριος Μπόντες για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, το 2008 ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζή ε, εξήγηλε την Ένωση για τη Μεσόγειο. Η Ένωση αυτή θα έδινε λέει νέα ορμή, νέο στόχο στις ευρωπαϊκές προσπάθειες και στους ευρωπαϊκούς στόχους που θα βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση κοινών αξιών όπως είναι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η καλή διοίκηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διερωτώ με, πώς είναι δυνατόν να μιλάει κανείς για κοινέ αξίες σε μια χώρα όπως τη Μαυριτανία, που δεν υπάρχει ανεξιθρησκεία ε, και το Ισλάμ ε, πάνω από ε, χίλια χρόνια κυριαρχεί. και άλλες χώρε, η Συρία α πούμε, που υποτίθεται ότι είναι σοσιαλιστικό κράτος και μονοκομματικό, είναι ε, δικτατορία. Τι γίνεται με τη Δυτική Σαχάρα, τι γίνεται με την Τινησία που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πού είναι ε, οι αρχές και οι αξίες, δεν έχω και χρόνο να τα πω. Ε, θέλουμε ε, καλή, συνεργασία, θέλουμε ελεύθερο εμπόριο με κάποιες χώρες και ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εκατέρωθεν της Μεσογείου. Αυτό θέλουμε να προωθήσουμε. Αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Ακόμα περισσότερο Ισλάμ θα εισάγουμε στην Ευρώπη πριν γίνει αυτό πραγματικότητα θα πρέπει να σταματήσουμε την προσπάθεια αυτή. Από το 1995 ονειρευόμαστε για τη Μεσόγειο με τη διακήρυξη της Βαρκελόνης. Και το 2005 τι έγινε. Τα σχέδια αυτά και τα έργα τα πληρώνουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και κάναμε μια τρύπα στο νερό. Σταματήστε αυτή την πατάληση διασπάτηση κονδυλίων και να ονειρεύεστε. Εγώ σέβομαι τον κύριο Αλμπερτίνη και τη θέση του που είναι θαραλέα και υποστηρίζεται και από την ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γιακολίνο, για 1,5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ευρωμεσογειακή Περιφέρεια αποτελεί μια στρατηγική περιοχή για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θεμελιώδη θέματα όπως το περιβάλλον, θρησκευτικέ αξίες, πολιτισμός, υποδομές, γεωργία, ενέργεια, ασφάλεια, μεταναστευτικές ροές χωρίς την υπεύθυνη συμβολή των τρίτων χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο στο ένα πλαίσιο συνεργασίας βέβαια το οποίο χρειάζεται ακόμα να διανύσει πολύ δρόμο. Από τη Βαρκελόνη, Βαρκελόνη και πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεσμευτεί περισσότερο στη διαδικασία ανανέωσης και επαλήθευσης των μεμονωμένων συμφωνιών σύνδεσης με τις τρίτες χώρες της Μεσογείου. Θα πρέπει να χρηματοδοτήσει τα μεγάλα στρατηγικά έργα για τις υποδομές και για τα λιμάνια. Και θα πρέπει όλα αυτά να παρακολουθηθούν ε, στεναρά. Το ε, ίδιο και για τη γεωργία, για να εγγυηθούμε την βιώσιμη ανάπτυξη και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορά όσο γίνεται πιο ομοιογενέ. Ευχόμαστε λοιπόν, θα θέλαμε λοιπόν την ενίσχυση του ρόλου της governance, τη διακυβέρνησης τη Ένωση για τις ευρωμεσογειακές χώρες για να επιβεβαιωθεί η αρχή της συνεργασίας που αντιπροσωπεύει πολιτική επιτυχία, επιχειρηματική ε, επιτυχία μέσα σε ένα βελτιωμένο πλαίσιο προστασία. και επίσης να προ να πω στην κυρία Μπεναράμπ ότι δεν είναι σωστό να επιτίθεται στο συνάδελφο Αλμπερτίν τη απουσία του για να μπορέσει και αυτός να υπερασπιστεί τον εαυτό του που είναι χαρακτηριστικό σε κάθε δημοκρατικά εκλεγμένη συνέλευση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντσέρη είναι ο επόμενος. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω πως ε, επιτελούμε ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά με την έγκριση αυτής της έκθεσης. Είναι πολύ χρήσιμη και εν ώψη τη διάσκεψη κορυφή τη 7η Ιουνίου στη Βαρκελόνη. Διάσκεψη κορυφή που, όπω γνωρίζουμε, προβλέπεται δύσκολη λόγω του μπλοκαρίσματο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ισραηλινού και Παλαιστινίου και λόγω μια αβεβαιότητα όσον αφορά την ορισμό τη διοικητική ε, δομής της νέας, της νέας γραμματείας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως οι συγκρούσεις δεν πρέπει να παρεμποδίσουν τη δυνατότητα συγκεκριμένης προόδου σε τομεακές συνεργασίες και πολυμερείς συνεργασίες. Και θα πρέπει επίσης να θυμίσουμε ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει με πλήρης επιτυχία της Ένωσης για τη Μεσόγειο χωρίς την επίλυση αυτών των διενέξεων. Και όλα αυτά περνούν μέσα από μια πολιτική σαφή δέσμευση ισχυρή που θα προέλθει από τη Βαρκελόνη. Νέα θεσμικά όργανα όργανα που θα μπορούν να λειτουργήσουν και να απελευθερώσουν τα απαραίτητα κονδύλια για την ε, ολοκλήρωση των μεγάλων προγραμμάτων που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι έχει δικά τη συμφέροντα προς τον Νότο για να μπορέσει να βρει λύσεις ε, στα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τώρα την νότια οχθή της Μεσογείου. Ευχαριστώ κύριο Ρινάλντι. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εδώ και χρόνια καταγράφουμε ένα σωρό κόσμο που προσπαθεί με, μικρά σκάφη να περάσει την Μεσόγειο. 4.200 άτομα έχουν ε, πνιγεί έτσι. Στη Λαπεντούζα. το παλιό κημητήριο εθελοντικά ε, ε, ενταφιάζει κάθε σώμα το οποίο βρίσκεται με έναν απλό σταυρό και ένα λουλουδάκι όλοι αυτοί οι πολίτες ενεργούν για τη δική μας, ε, δικό μας λογαριασμό και ανταποκρίνονται έτσι στη δική μας πολιτική αποτυχία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια άλλη αρχιτεκτονική πολιτική διαφορετική από αυτή της Ιταλικής ε, κυβέρνησης. Προσθέτουμε μόνο έτσι στην απελπισία αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει δηλαδή η, Ευρωπαϊκή, η Ένωση την Ευρώπη να ανακαλύψει μια νέα ένα νέο ανθρωπισμό. Δεν έχουμε χρόνο. Πάνω από το μισό πληθυσμό του, από το Μαρόκο μέχρι την Τουρκία, είναι κάτω των 18 ετών. Άρα λοιπόν η Μεσόγειος ε, ε, έχει προορισμό να αλλάξει πολύ πολύ γρήγορα. Επόμενος ο μιλητής κ. Χατζηγεωργίου. Παρακαλώ δύο λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπεγιόν για τη δουλειά που έχει φέρει σε πέρας η έκθεση καλεί τι κυβερνήσει των κρατών μελών της Ένωση για τη μεσόγειο να εγκαθιδρύσουν έναν ανοιχτό διάλογο στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και της αλληλοκατανόησης με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και αυτό είναι κάτι που στηρίζομαι. την ίδια ώρα όμως δεν περιλαμβάνει καμιά ουσιαστική πρόταση για αντιμετώπιση των υφιστάμενων πολιτικών προβλημάτων που ταλανίζουν την περιοχή κατανοώ τη λογική του συναδέλφου κυρίου Πελιών που υπάρχει πίσω από αυτό το λεχτικό και που μάλλον θεωρείται υποβοηθητική στο ξεκίνημα της ένωσης. από την άλλη όμως το να κάνουμε τους τυφλούς και να προσποιούμαστε ότι δεν τρέχει τίποτα στη γάζα για παράδειγμα είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος που μας κάνει να ζούμε με την σκόνη πάνω από τα προβλήματα. φοβούμαι αγαπητοί συνάδελφοι ότι στην ευρωπαϊκή ένωση σιγά σιγά εκπαιδευόμαστε να ζούμε με τα προβλήματα αντί να τα λύουμε. πρέπει να μπαίνουμε πιο δυναμικά πάνω στα ουσιώδη ζητήματα που μας απασχολούν. απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην ανάγκη όπως το ισραήλ προχωρήσει σε μια άμεση δίκαιη και βιώσιμη διευθέτηση του παλαιστινιακού. απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην ανάγκη όπως η τουρκία δείξει τον αναγκαίο σεβασμό προς όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη της ένωσης για τη μεσόγειο η υπόδειξη του χρέου για απόσυρση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων από ένα κράτο μέλο είναι μια αναγκαία πράξη σεβασμού προ το μίνιμουμ θα έλεγα μια Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. η Μεσόγειο αγαπητοί φίλοι βρέχει μερικέ χιλιάδε πόλεις και χωριά διαφορετικέ κουλτούρε με ενοποιητικά στοιχεία γύρω από την ίδια θάλασσα για δέκα και πλέον χιλιάδε χρόνια. μόνο μια πόλη όμω από αυτέ τι χιλιάδε πόλει και χωριά που βρίσκονται στι παραλίε τη μεσογείου μόνο μια πόλη είναι ακατοίκητη. αντί ανθρώπων την κατοικούν ποντίκια σαύρες και φίδια. τα σπίτια των ανθρώπων μαζί με τις μνήμες έχουν διαβρωθεί. μένουν μόνο τα όνειρα χιλιάδων ανθρώπων πολλοί από τους οποίους έχουν πεθάνει πρόσφυγες. δεν θα είναι το ελάχιστο που χρωστούμε στους ζωντανούς να επιστραφεί η πόλη τους αμοχώστους τους κατοίκους της. έπρεπε αυτό να ήταν βασική απέτηση της έκθεσης. Mm, για την ένωση για τη μεσόγειο γιατί δουλεύουμε για την ένωση για τη μεσόγειο και όχι για τη διχοτόμηση στη μεσόγειο. ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπάτμ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας συνήθως δεν σημαίνουν τίποτα, δεν καταλήγουν πουθενά. Μπορούν όμως και να εκφράσουν την πολιτική θέληση του Κοινοβουλίου. Η έκθεση αυτή προτείνει δημιουργία μιας ένωσης 17 μη ενωσιακών χωρών με κοινέ συναντήσεις των βουλών, γραμματεία και αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα φιλόδοξο. Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου προγράμματος θα σήμαινε εκατομμύρια που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι και οι φορολογούμενες. Από πού θα προέρθουν τα χρήματα αυτά, αυτό δεν μας το λένε. Είναι όλα φαντασίες χωρίς καθόλου πραγματικότητα. Πρέπει πριν την καταδικάσουμε όμως να θυμηθούμε ότι η Ένωση έχει τη δυνατότητα να υπογράφει τέτοιου είδους συμβάσεις βάσει της ε, συνθήκης Λισαβόνας. Έτσι ώστε οι χώρες αυτές εν καιρό το δένδυ να απορροφηθούν και αυτές στην Ένωση. Αυτό στοχεύει η έκθεση. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Μέλτσερ παρακαλώ. Πριν από δύο χρόνια και ιδρύθηκε Ένωση για τη Μεσόγειο και υποτίθεται ότι θα ε, έπρεπε να συνδεθεί με τη διαδικασία της Βαρκελόνης για πιο στενή σύνδεση των κρατών της Μεσογείου με την Ένωση. Προφανώς όμως λόγω της σύγκρουση μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραήλ έχει αποτελματωθεί αυτή η υπόθεση. Ε, γνωρίζουμε ότι έχουμε συμφωνίες σύνδεσης και με το Ισραήλ και μόνο στη Γάζα δίνουμε 440 εκατομμύρια βοήθεια. Και διερωτώνται οι ε, φορολογούμενοι στην Ευρώπη γιατί ε, θα πρέπει να στέλνουμε τόσα λεφτά στη Γάζα αφού ξανά και ξανά τα βομβαρδίζουν και τα ισοπεδώνουν χωρίς συνέπειες. Και ε, τελικά δεν αποκλείεται ότι και η Χαμάς επωφελείται από τα χρήματα αυτά. Δεν κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμφανιστεί ε, διαμεσολαβητής ανεξάρτητος στη Γάζα. Και έχουμε τώρα τη ε, Βαρκελόνη που ε, δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή η διαδικασία στην επίλυση της διαφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε την κατάσταση σωστά και ενδεχομένως να την διακόψουμε, να την αναστείλουμε. Τι να τα κάνουμε. Αυτά είναι θέματα κύρους και στέλνουμε εκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποντής παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Ah, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της Βαρκελόνης, η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι μια ευκαιρία για την ανάπτυξη σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου. Όπως το τονίζει η εξαιρετική έκθεση του Βικεντίου Πεγιών, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ούτε το δυναμικό αυτής της περιοχής ούτε και τον κίνδυνο που μπορεί να εμπεριέχει. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι από τους βομβαρδισμούς της Γάζης και την συνέχιση του επικισμού των Παλαιστινιακών εδαφών η Ένωση για τη Μεσόγειο βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η πολιτική της πτυχή έχει τελείως παγώσει και δεν είμαστε καν βέβαιοι ότι η διάσκεψη του Ιουνίου στη Βαρκελόνη θα γίνει πράγματι. Δεν θα με ξέπλυσε αν μαθαίναμε τις επόμενες μέρες ότι ακυρώνεται ή αναβάλλεται. Δεν πρέπει όμως να παρετηθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της στην, για την εξερεύνηση μιας πολιτικής λύσης. Δεν μπορούμε να αφήσουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες το μονοπόλιο της πολιτικής διαχείρισης της κρίσης της περιοχής αυτής που είναι δική μας εφόσον βέβαια δεχτούμε να συμφωνισφάρουμε και στην ανάπτυξή της. Η σταθερότητα στη Μεσόγειο ε, είναι κάτι από το οποίο εξαρτάται και η δική μας ασφάλεια και γι' αυτό η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι το καλύτερο εργαλείο που, μπορούμε να, που διαθέτουμε για να τη διασφαλίσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόπα. Χαρώ τον εισηγητή για την πληρέστατη έκθεσή του η ένωση για τη μεσόγειο μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας ισορροπημένης ευρωμεσογειακής σχέσης καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις χώρες της περιοχής. η μεσόγειος πρέπει να είναι μια περιοχή ειρήνης σταθερότητας και ασφάλειας όπου οι δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται πλήρως σεβαστά. οι κοινωνικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ των μεσογειακών χωρών είναι δεδομένες. το στίχημα είναι ακόμα μεγαλύτερο λόγω της οικονομικής κρίσης αφορά την ουσιαστική προσέγγιση της ένωσης με τις μεσογειακές χώρες μέσω της ανάπτυξης της συνεργασίας και του εμπορίου. η ενεργειακή ασφάλεια η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής το θαλάσσιο περιβάλλον είναι επίσης επιβεβλημένα πεδία στενής συνεργασίας. η ένωση για τη μεσόγειο δεν είναι φυσικά το πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές συγκρούσεις. όμως η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας ο πολιτικός διάλογος και η κοινή προσπάθεια σε συγκεκριμένους στόχου συμβάλλουν καθοριστικά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνη κάτι που είναι αναγκαίο για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων. για να γίνουν όμω όλα αυτά και να πετύχει η ένωση για τη μεσόγειο χρειάζονται απαραίτητα τα κατάλληλα δημοσιονομικά μέσα και αυτή τη φορά δεν πρέπει να ολιγορήσουμε. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Ε, ήμουνα σε άλλη επιτροπή σε, στο Προεδρείο και καθυστέρησα. Ευχαριστώ. Ε, σωστά η έκθεση Πεγιό στην παράγραφο 5 σημειώνει την ανάγκη ε, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στην Ισραηλινο-Αραβική διένεξη. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουν όσο μπορούν προς την κατεύθυνση αυτή. Κατά την άποψή μου, και επειδή είμαι και πρόεδρος της αντιπροσωπής για το Ισραήλ, πραγματικά θέλω να υποστηρίξω αυτό. Αλλά για να πετύχει αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να ισχύουν οι δύο όροι και προϋποθέσεις. Πρώτον, να πούμε ξεκάθαρα ότι θα υπάρχουν δύο κράτη. Δύο κράτη. Ένα, ένα κράτος εβραϊκό, το Ισραήλ, και ένα κράτος παλαιστινιακό. Να το πούμε αυτό. Και δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινή προσπάθεια για να ε, καταστραφεί αυτό το ενδυμικό δεινό εκεί που είναι ο αντισημιτισμός. Μόνο έτσι θα προχωρήσει η προσπάθεια αυτή και χρειάζεται κοινή προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή. Ο κύριος Μιγιάν Μον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια εισαγωγική διευκρίνηση. Κάποιο από το Συμβούλιο δεν θα έπρεπε να είναι εδώ από την Προεδρία ή από την Ένωση για τη Μεσόγειο, από την γαλλική πλευρά και να μιλήσει. Λυπάμαι πάρα πολύ για την απουσία αυτή. Κυρίε και κύριοι, για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό η πιο κοντινή γειτονία τη να είναι χώρο ασφάλεια, δικαιοσύνη, εφημερία και ελευθερία. Αυτό θα πρέπει να είναι στόχο και τη Ένωση για τη Μεσόγειο που ελπίζω η δεύτερη σύνοδο κορυφή να διεξαχθεί τον επόμενο μήνα. Ε, χαίρομαι και συγχαίρω τον κύριο Πεγιόν και για το ανοιχτό και επικοδομητικό του πνεύμα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και με την νότια όχθη τη Μεσογείου έχουμε πολλέ διαφορέ πολιτικέ, κοινωνικέ, οικονομικέ, ε, εθνικές, πολιτισμικέ κτλ. Και έχουμε σοβαρέ ανεπάρκειε στα κράτη αυτά που είναι οι γείτονέ μα. Ε, Στενό διάλογο, στενή συνεργασία για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Μεγάλα έργα από κοινού και ε, διμερέ σχέδιο για τι συμφωνίε σύνδεση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ απαραίτητα για να ενισχυθεί η συνεργασία των όχθων και να καταφέρουμε να μειωθούν οι διαφορέ. Θα πρέπει όμω και οι γείτονέ μα να κάνουν μεταρρυθμίσει. Δεν θα, πρέπει να είναι επιλογή η ακινησία και η πράξη. Θα ήθελα να τονίσω τα εξή ακόμα. Πρώτον, το συντομότερο να είναι πλήρω λειτουργική γραμματεία στη Βαρκελόνη. Δεύτερον, και αυτό συνδέεται στενά με το προηγούμενο. Η Ένωση για τη Μεσόγειο δεν μπορεί να είναι όμοιρο των ε, διενέξεων και των σειράξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να δώσει τη λύση, ούτε πρέπει να μπλοκάρεται από αυτέ τι εξελίξει. Και τέλο, ε, Πρόεδρε, η Ένωση για τη Μεσόγειο επίσης θα πρέπει να δώσει κατά προτεραιότητα προσοχή στο λεγόμενο τέταρτο άρθρο της συνεργασίας που είναι τα μεταναστευτικά ρεύματα, ασφάλεια, κοινωνική ένταξη και δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω να ζητήσω συγγνώμη ότι, γιατί οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα το πρωί γιατί είναι πέμπτη το πρωί και αρχικά είχε προγραμματιστεί η συζήτηση αυτή για τη Δευτέρα. Αυτή είναι η δικαιολογία του Συμβουλίου. Διαδικαστικό κύριο Πόσελτ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω στον τριμερή διάλογο να υποβάλλεται ε, το αίτημα να είναι πάντα παρόν το Συμβούλιο την Πέμπτη το πρωί. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, δεν θα σας πω τώρα χώρες, ε, και μάλιστα και Πέμπτη απόγευμα. Και θεωρώ πραγματικά ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι παρόν κατά το μεγαλύτερο τμήμα της Ολομέλειας. Ευχαριστώ, θα το κάνω, λέει ο Πρόεδρος. Προσπάθησα να εξηγήσω μόνο την απουσία του Συμβουλίου, ε, τι μας είπαν. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι η ομιλήτρια κυρία Ανδρέας Μπαρέα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τεσανέζα από την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου για τη συνεργασία μας. Περισσότερο από ποτέ σήμερα είναι απαραίτητη η Ένωση για τη Μεσόγειο, ενίσχυση των μεγάλων έργων και η θεσμική ανάπτυξη. Περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να βρεθούν λύσεις για να βγούμε από την κρίση ε, για την έρευνα, για την κλιματική αλλαγή, για το νερό, για την ενέργεια, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε καλές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ε, με μέτρα βράχη πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, ε, ε, άρση των τελωνιακών φραγμών, διάνοιξη αγορών βορρά νότου και νότου νότου. Η Ισπανική Προεδρία θα δώσει την ευκαιρία στη Βαρκελόνη για μια νέα δέσμευση, για μια νέα κατάσταση και για ένα νέο στίχημα εκδημοκρατισμού, οικονομικών λύσεων και κοινωνικών λύσεων η σύνοδο κορυφή τη Βαρκελόνη μπορεί να μα φέρει σε ηγετική θέση στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα η συνεργασία ανάμεσα οι επαφέ μάλλον ανάμεσα στου μεσογειακού λαού ε, εκδηλώνονται μέσω του εποχιακού φαινομένου τη μετανάστευση. Αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι μεταναστευτικέ ροέ οδηγούν και προκαλούν προβλήματα στο ανθρώπινο, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο. Ποιες ποιο θα είναι δηλαδή το ίδιο το μέλλον των δυο όχθεων της Μεσογείου. Η εγκύτητα των λαών Μεσογείου εκδηλώνεται και μέσα στο πλαίσιο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω των εμπορικών συναλλαγών και ανάμεσα στις, και μέσα στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Είμαστε ριζωμένοι σε αυτή την περιοχή και θα πρέπει να αποφύγουμε η Ένωση για τη Μεσόγειο να πέσει στις αντιφάσεις της Βαρκελόνης. Πόσα σφάλματα, πόσες φορές σκεφτήκαμε ότι θα κάνουμε βήματα εμπρό, ενώ στην ουσία πιστοδρομούσαμε. Αυτό που θα πρέπει να εγκατασταθεί καταρχήν είναι ένας κοινωνικός, πολιτιστικός, ανθρώπινος διάλογος που θα έχει ως προϋπόθεση την αμοιβαία κατανόηση και την προώθηση των καλών αξιών που ε, θεμελιώνουν τον πολιτισμό μας. Όμως αυτός ο παράγοντας, ε, ο αδιαμφισβήτητος, ε, στην ουσία βασίζεται καταρχήν στη συνεργασία την οικονομική. Ο πολλαπλασιασμός των σχέσεων και των συναλλαγών ευνοεί την επέκταση των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων, οι οποίε δεν είναι ισόρροπε ανάμεσα στα μέρη. Επιπλέον, σε πολιτικό επίπεδο, είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε με μια κατάπαυστη ε, ε, αναζήτηση διαλόγου που αφορά την πολιτική ασφάλεια, ώστε να υπάρξουν όλο ένα και πιο στενέ σχέσει ανάμεσα στι ε, ενδιαφερόμενε χώρε. Παρακαλώ, συνάδελφοι, να κρατάτε το χρόνο σα, γιατί στι 12 έχουμε ψηφοφορίε. Κύριε Πυρίλο, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η διάσκεψη κορυφή των ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 7 και 8 Ιουνίου στη Βαρκελόνη αναμφίβολα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη συγκεκριμένη δρομολόγηση της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Είναι μια εξαιρετική ε, περίσταση για να δημιουργηθούν οι βάσεις για μια αληθινή και πιο ισχυρή συνεργασία υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας. Ακριβώς γι' αυτό είναι απαραίτητο αυτή η ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να οικοδομηθεί μια στρατηγική ανάπτυξη και να φτάσουμε στην ολοκλήρωση προγραμμάτων που θα είναι σε θέση να στηρίξουν ολόκληρη την περιοχή και να ευνοήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Ελπίζω πως από την ε, ε, συνάντηση αυτή θα προκύψουν πρωτοβουλίε όπως οι ε, ειρηνευτικές αλλά και μέσα για την δημιουργία ενός μέσου για την ενέργεια. Επίσης, προώθηση της ενέργειας και της έρευνας συγγνώμη, και της ανάπτυξης της τεχνολογίας ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων που συχνά είναι πολύ αδύναμες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς. Είμαι επεπισμένος πως η συμβολή της Ένωσης θα ενισχύσει η συμβολή της, Ευρωπα... Ε, ε, της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα ενισχύσει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση για την Ένωση για τη Μεσόγειο απαιτεί αυτή τη στιγμή μια αποτίμηση και αξιολόγηση των προοπτικών της. Γι' αυτό θεωρώ ότι η έκθεση του κυρίου Βενσάν Πεγιό ε, είναι τελείως επίκαιρη και θα ήθελα όπως και οι άλλοι συνάδελφοι να τον συγχαρώ και εγώ. Η διάσκεψη του Ιουνίου της Βαρκελόνης πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία όπου το Κοινοβούλιο να επαναλάβει τη δέσμευσή του να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή για την ανάπτυξη της περιοχής αυτής που είναι στο σταυροδρόμι όλων των εξελίξεων και έχει πολύ σοβαρή γεωστρατηγική θέση. Άκουσα τις αμφιβολίες του κύριου Μποντής ως προς τη δυνατότητα διοργάνωσης της διάσκεψης αυτής. Ελπίζω να γίνουν όλες οι προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί και να αποτελέσει μια ευκαιρία όχι μόνο ανάλυσης αλλά και θεσμικής επιτυχίας, διότι η Ένωση αυτή πρέπει να ξεπεράσει τους πολιτι... και τα πολιτικά προβλήματα και να καταλήξει σε ένα στρατηγικό πρόγραμμα που να βοηθήσει και τις δύο όχθες. Η αξιοπιστία της εξαρτάται από τη δυνατότητά της να δράσει και γι' αυτό χρειάζεται επαρκής χρηματοδότηση ώστε το όραμα αυτό να επιτύχει και η γραμματεία να λειτουργήσει πραγματικά με συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων ώστε να υπάρχει και η απαραίτητη δημοκρατική νομιμότης. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα περάσουμε στην οφθαλμοθυρία. Ένα λεπτό ο καθένας και η καθεμία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συμβολή στην πλήρη επιτυχία τη επόμενη διάσκεψη κορυφή τη Βαρκελόνη. Μετά από δύο χρόνια τελμάτωση από την διάσκεψη του Παρισιού του 2008, είναι πολύ οι στόχοι, του θυμήσαμε και σήμερα, κατά πολέμηση τη λαθρομετανάστευση, πολέμηση τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά υπάρχει και μια σημαντική οικονομική πτυχή. Η Μεσόγειος ε, προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ε, με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να στηριχθεί το ηλιακό πρόγραμμα για την Μεσόγειο και πρωτοβουλίε βιομηχανικέ όπω η Desert Pack που συμμετέχουν εταιρείε και τα πανεπιστήμια με στόχο συγκεκριμένα προγράμματα συνεργασία. Ε, η ειρηνευτική διαδικασία που είναι προτεραιότητα θα πρέπει να συνοδευτεί από μια διαδικασία οικονομική ανάπτυξη ακριβώ για να εγγυηθούμε αυτή την συνοχή, την, την κοινωνική συνοχή που είναι απαραίτητη για να βοηθήσει στην υπέρβαση των συγκρούσεων. Ευχαριστώ. Η κυρία Σανάλοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι πολύ τολμηρό ε, βήμα. Θα πρέπει να δούμε αν είμαστε πρόθυμοι να συνδυάσουμε τις διαφορετικές μας παραδόσεις ε, ε, ε, τις, όλες τις διαφορές που έχουμε, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι η ισότητα των φίλων στην κοινωνία. Είναι πολύ ευαίσθητο και κομβικό θέμα ακριβώς σε αυτή την περιοχή και η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ και με αυτό το θέμα. Όχι μόνο επειδή εμείς εδώ ε, έχουμε τη διάσκεψη του Μαρακές του 2009 που έχει αναλάβει την ε, ευθύνη και την αποστολή να υποστηρίξει την ισότητα των φίλων, να υποστηρίξει συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική ζωή και να καταπολεμήσει τη βία κατά των γυναικών. Αυτό ε, θα ήταν μεγάλη πρόοδος για όλη την περιοχή και θα ήταν κέρδος και μόνο είναι διαφορετικές οι παραδόσεις, επαναλαμβάνω, διαφορετικά τα δεδομένα, διαφορετικά εμπόδια ε, που δεν βοηθούν στην ανάπτυξη περιοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει ε, το πρόγραμμα τη της Ένωσης για τη Μεσόγειο από πολιτικής και από οικονομικής άποψη. Στις 7 Ιουνίου στη Βαρκελόνη θα γίνει η διάσκεψη κορυφής των 43 επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης για τη Μεσόγειο και όπως και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ευχηθούμε σε αυτό το ραντεβού αυτό το ραντεβού να είναι επιτυχές για την Ένωση, για τη Μεσόγειο και για την υλοποίηση των προγραμμάτων Ω και και συζητητής ε, για την χρωμοδότηση στην έκθεση ΙΤΡΕ, εγώ έχω υπογραμμίσει σημεία που είναι θεωρώ σημαντικά, όπω η υλοποίηση μια ε, ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με τι χώρε τη Μεσογείου, τη συμμετοχή του τομέα τη έρευνα ε, και της παιδείας, ενάπτυξη της ευρεία ζώνης, επίσης βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πω ότι αυτές αντιπροσωπεύουν ήδη έναν από τους στρατηγικούς τομείς. Τα μεγάλα προγράμματα θα πρέπει να κατάλληλα να υποστηριχτούν από τα ευρωπαϊκά και διεθνή οικονομικά ε, όργανα για να μπορέσουμε να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι Ευρωπαίοι partner. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Πρόεδρε, η πρόταση του Πρόεδρου Σαρκόζη για την Ένωση για τη Μεσογείο αποτέλεσε το αποκορύφωμα για την ε, Γαλλική Προεδρία. Έκτοτε φαίνεται να έχασε τη λάμψη του, γιατί ούτω ή άλλω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προχωρήσει πολύ για την, Ευρωπαϊκή, για την πολιτική γυτνίαση ε, με του νότιου γείτονέ τη. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι βλέπουν ωστόσο ότι γίνεται μια επικάλυψη προσπαθειών και μια κατασπατάληση των πόρων. Όποια και αν είναι το μέλλον της Ένωση για τη Μεσόγειο, στην διάσκεψη κορυφής της 7 Ιουνίου δεν πρέπει να ε, ε, ε, επιτρέψουμε να μείνει πίσω η ανατολική διάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. έχει καθυστερήσει η δημιουργία της συνέλευσης, ιδιαίτερα λόγω της, ε, Λευκορωσία, λόγω της Λευκορωσίας. Τώρα, ο πρόεδρος Αλμπερτίνη αποφάσισε να μην συμμετέχει. Συζητήθηκε και στην ε, ε, διάσκεψη των Προέδρων σήμερα το πρωί. Πάντως, οποιαδήποτε πρόταση για απαραίτηση, εμείς θα, την, αντισταθούμε. Ο κύριος Βερμπάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και χιλιετίες ε, είναι το λίκνο του πολιτισμού μας η Μεσόγειος και η κινητήρια δύναμή μας. Και καλωσορίζουμε την Ένωση. Είναι όμως και μια γέφυρα για χαλήνο τη μετανάστευση προς την Ευρώπη και μάλιστα η λαθρομετανάστευση είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και έχουμε έξι στρατηγικούς τομείς που το καταπολεμούν αυτό αλλά μόνο με κοινή ε, συνεργασία των χωρών της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής μπορούμε να σταματήσουμε αυτά τα ρεύματα ή να τα ελέγξουμε αν μη τι άλλο. Μόνο έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό στην πηγή. Εκεί θα πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση καταπολεμώντας την ένδια γιατί είναι και λαθρεμπόριο, είναι οργανωμένο έγκλημα αυτό που γίνεται εκεί. Υποτιθέμενη χρυσή Ευρώπη ε, δεν είναι το Ελντοράντο, δεν έχει δουλειά για όλους, στέγη για όλους, άσυλο για όλους. Γιατί τελικά έχουμε και επαναπροωθήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλτασάρη έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Παρά τη δημιουργία της Ένωσης και την διάσκεψη κορυφής εξακολουθεί να λείπει ένα σαφή ορισμό τη μεσογειακή πολιτική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο, μακρόπνο όραμα για την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση τη περιοχή. Και ωστόσο το δυναμικό τη Μεσογείου είναι τεράστιο. Εν τρίτο του διεθνού τη διεθνού ναυσιπλοεία γίνεται στις, στα νερά τη Μεσογείου, από την Κίνα, από την Ασία, από τι Ευρωπαϊκέ χώρε, από την Ινδία και μέσω από το ΣΟΕΣ φτάνει στα υδατά μα. Οι παρόχθες χώρε ε, από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Αφρική είναι αναπτυσσόμενε, είναι ήδη προηγμένε ε, στην ανάπτυξή του. Είναι πολύ σημαντική τομή ε, συνεργασία μαζί. Γι' αυτό και θα πρέπει να θεσπίσουμε καλύτερα και να ορίσουμε καλύτερα τι δομέ συνεργασία σε δίνοντας στη Γραμματεία της Ένωσης για την Ευρώπη τα απαραίτητα μέσα και τα κριτήρια προσχώρησης και υλοποίησης των προγραμμάτων. Ορισμένα σημεία κλειδιά, γεωργία, μεταφορές, θαλάσσια αυτοκινητόδρομοι, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακό πρόγραμμα, έλεγε ο Πολ Μωράν που ήταν διπλωμάτης και συγγραφέας Γάλλος, έλεγε πως η Μεσόγειος είναι ο πολιτισμός του νερού και της ε, ερήμου. Η κυρία Ντότ. Uh, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω για το πώς θα μπορέσει ο φορολογούμενος και η φορολογούμενη να πληρώσει για τα έξοδα λειτουργίας αυτής της γραμματείας αλλά θα ήθελα να σας εκφράσω την άποψή μου ότι χωρίς αμφιβολία η σταθερότητα στη Μεσόγειο είναι σαφώς κάτι θετικό για την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό σημαίνει και ευθύνη της Ένωσης αν θέλει να βοηθήσει τις χώρες της Μεσογείου, της Νότιας Όχθης Μεσογείου να αναπτυχθούν πολιτικά και οικονομικά. Και θα τονίσω μία πτυχή, δηλαδή την απόρριψη χιλιάδων τόνων σπόρου πατάτας στη θάλασσα από τις μαροκινές αρχές στην Ιρλανδία. Πριν φύγουν από την Ιρλανδία Είχαν θεωρήσει, είχαμε θεωρήσει ότι ε, ε, εφήρμοζαν τους ισχύοντες κανόνες αλλά μόλις φύγανε πέταξαν τους σπόρους στη θάλασσα. Θα ήθελα να τονίσω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευθύνη από όσους θέλουν να ωφεληθούν από τέτοιου σχέδια. Ευχαριστώ. Επίτροπος Φίλε έχει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much, uh, Madam uh, President. It has been a good and inspiring uh, Ευχαριστώ. Α, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, δεν ήμουν έτοιμος ψυχολογικά. λοιπόν. Ναι, ήσασταν πολύ γρήγορος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πολύ καλή αυτή η συζήτηση και διαφανής μάλιστα, συζήτηση διαφανής. Πολλοί έχουν πει δικαίω ότι χάσαμε πολύ καιρό, ιδίω ω προ την διοργάνωση τη γραμματεία. Θα το πω σε λίγο αυτό. Ακόμη αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, όπως το πώς θα διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε γίνει για τη διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή δεν θα πάρει σαν όμοιρο την Ένωση για τη Μεσόγειο. Δεν θα γίνει εκβιασμός δηλαδή ότι θα διοργανωθεί πράγματι η διάσκεψη και θα δημιουργήσει μια νέα ορμή Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα επιληθεί και το πρόβλημα της διακυβερνητικής έναντι της ενωσιακής αντιμετώπισης. Πέντε σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτον, συνεργαστήκαμε με την Ισπανική Προεδρία για πολλούς μήνες και μαζί ε, ιδρύσαμε τη γραμματεία την 1η Μαρτίου και έκανε πολλές προσπάθειες η Ισπανική Προεδρία ώστε να διοργανωθεί πράγματι η διάσκεψη του Ιουνίου. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό η γραμματεία να χρηματοδοτηθεί επαρκώς. Παραδείγματος χάρη από την Κομισιόν να στείλει έναν εμπειρογνώμονα που να διασφαλίζει ότι υπάρχει συμβατότης μεταξύ του προγράμματός της και των ενωσιακών στόχων να μην είναι τεράστια αλλά να έχει και επαρκή επάνδρωση ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη και πολλαπλασιασμός των προγραμμάτων. Επίσης σημαντικό θα ήταν να πούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι πολλές τομεακές συναντήσεις διοργανώνονται. Την επόμενη εβδομάδα ε, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών, την μεθεπόμενη Υπουργή Γεωργίας στο Κάιρο. Η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τμήμα της πολιτικής μας καλής γειτονίας αλλά το κυριότερο στοιχείο των σχέσεών μας είναι διμερές. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερη δέσμευση από όλους μας τους εταίρους και ως προς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κινητικότητας που είναι και αυτή κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και συμφωνώ με όσους ζήτησαν να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας και των χωρών της Μεσογείου. Τέλος, η επόμενη ευκαιρία για να κάνουμε την προσπάθεια αυτή θα είναι η αξιολόγηση των πολυμερών και διμερών σχέσεων που έχουμε με τις χώρες αυτές. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Ο εισηγητής τώρα ο κύριος Βικέντιος Πεγιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε πίτροπε. Καταρχήν, τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, τους σεβαστήκαμε όλους και ιδιαίτερα τα θύματα. Θεωρήσαμε ότι η αγανάκτηση όμως δεν αρκεί για να δημιουργήσει πολιτικό πρόγραμμα. Δεν αρνούμε τις διενέξεις που υπάρχουν ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Παλαιστίνη, ούτε στη Δυτική Σαχάρα. Αλλά είμαστε σοβαροί. Στην εξωτερική πολιτική, ε, στην ΚΕΠΑ, στις διάφορες επαφές που έχουμε είπε κανείς ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο πρέπει να λύσει αυτά τα πράγματα ούτε βοηθάει η σύγχυση στην αποτελεσματικότητα. Επίσης λυπούμε και εγώ για την απουσία του Συμβουλίου. Δεν είναι καλό δείγμα αυτό και δεν είναι καλό δείγμα όταν ακούμε ότι ε, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Έχει δίκιο ο Μποντής ότι η σύνοδος ε, της 7 η Ιουνίου διακυβεύεται ίδια. Το Κοινοβούλιο ανέλαβε τις ευθύνες του. Εκείνοι που οικοδόμησαν την Ευρώπη, την οικοδόμησαν ε, και με μεγάλο στένος και θέληση ε, και με συγκεκριμένη πολιτική βούληση, με τη στενή έννοια μετά από τους πολέμους που μας αιματοκύλησαν και μας δίχασαν. Η Ευρώπη διανύει αυτή τη στιγμή μια κρίση σημαντική και θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ανάπτυξης ε, και όχι αναδίπλωσης. Η αναδίπλωση ε, και η πάυση των ε, σχέσεων με το εξωτερικό σημαίνει αργό θάνατο. Η συλλογική εργασία αυτή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και εύχομαι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, πράγμα που δεν τους χαρακτηρίζει το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Πεγιό. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα ακολουθήσει στις 12. Επόμενο θέμα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, είναι η έκθεση του κυρίου Κύριλοφ με θέμα την αναγκαιότητα μια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Νότιο Κάφκασο. Ο εισηγητή έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Mr. President, dear Commissioner Fule... Κύριε Πίτροπε Φούλε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω